Iniziamo i nostri lavori che oggi non sono particolarmente gravosi. Io eh, comunicherò in primo luogo le raccomandazioni. Έχουμε πάρα πολλέ εργασίε. Θα ήθελα να σα πω ότι έχουν κάνει οι συντονιστέ. Και συνεχεία θα πρέπει να πάρουμε αποφάσει για την ακρόαση του αρμοδίου επιτρόπου για τα θέματά μας. θα πρέπει να αποφασίσουμε για τη δική μας συμμετοχή σε άλλες ε, ακροάσεις ενδεχομένως. Και συνεχεία θα ασχοληθούμε με το θέμα ΚΟΖΑΚ, την, ε, τους ειδικού ε, οργανισμούς των Εθνικών Κοινοβουλίων. θα έρθει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα ο Αντιπρόεδρος Σκοτ Μακμίλαν. Και στο τέλος θα πρέπει να μιλήσουμε για τις εκθέσεις εν γέννη, όχι αυτό το είπα. Αυτά. Θα ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις και τις συστάσεις από τους συντονιστές. Στις 19 Οκτωβρίου είχαμε την προηγούμενη συνεδρίασή μας. Εκεί αποφασίσαμε να μην εκπονήσουμε έκθεση για τη διαδικασία απαλλαγής ε, του προϋπολογισμού του 2008. Ενώ χθε, μετά την μακρά συνεδρίαση, η συνεδρίαση των συντονιστών έκανε τις εξής προτάσεις, άλλες προτάσεις. Διορισμός ενός ε, εισηγητή για τις εκθέσεις ε, για τις, της Οικονομικής Επιτροπής, για τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θεσμικά θέματα για την οικονομική εποπτεία. Μιλάμε για πέντε εκθέσεις και οι συντονιστές λένε να εκφραστούμε μέσω μιας έκθεσης, αλλά μέσω μίας, όχι μέσω πέντε. Ο το ΕΛΚ ζητάει να διορίσει τον ε, εισηγητή σε αυτή την έκθεση, τον έχει. Τώρα, για την έκθεση της Νομικής Επιτροπής, για την έκθεση πρωτοβουλίας της 16ης έκθεσης του Εθνομοθετή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι, φαίνεται ότι υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της νομικής επιτροπής για αυτό το θέμα. Αλλά επειδή στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας ζητείται να υπάρξει εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ένωσης και Εθνικών Κοινοβουλίων, ιδίως ό,τι αφορά τον έλεγχο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάτι που αφορά τη δική μας, τις δικές μας αρμοδιότητες, την δική μας εντολή, θα πρέπει και εμείς να είμαστε παρόντες. Στις 10, στις 10 του Νοεμβρίου βεβαίως θα συνεδριάσει η Νομική Επιτροπή και τότε θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει όντως να παρέμβουμε, αλλιώς θα παρετηθούμε. Θα δούμε λοιπόν τότε αν υπάρχουν αρμοδιότητες δικές μας. Το ΕΛΚ παρόλα αυτά ζητάει να διοριστεί ένας ε, αρμόδιος και ως συνήθως στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι και ένας βουλευτής υπεύθυνο για θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Προτείνουμε να διορίσουμε την Αντιπρόεδρο Γκουρμάη ως υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Εν συνεχεία, αποφασίστηκε να σας προτείνουμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας ε, ε, προβληματισμού, τον Φελίπε Γκονζάλες, ε, στην επόμενη συνεδρίαση ε, για τα θέματα προβληματισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, προτείνεται να δεχτούμε την εξή ιδέα, να εκπονήσουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την αθεώρηση των τρόπων διερεύνηση των ερευνητικών επιτροπών, των τρόπων εργασιών λοιπόν. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζήτησε να πάρει αυτή την έκθεση γιατί έχει και τρεις πόντους. Άλλος εισηγητής τώρα θα πρέπει να διοριστεί για την αναθεώρηση της ε, Συμφωνίας Πλαίσιο ε, Κομισιόν Κοινοβούλιο. Εδώ πάλι υπάρχει ένα αίτημα του ΕΛΚ, δύο πόντι, ε, δύο βαθμοί για αυτή την έκθεση. Επίσης εκπώνησε έκθεση πρωτοβουλία για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο τίθεται σχέση με την συνθήκη της Λισαβόνα. Είναι μια προαίρεση βεβαίω, όχι μια υποχρέωση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν και πώς θα προσχωρήσουμε στην ε, Ευρωπαϊκή αυτή σύμβαση. Ε, προτείνουμε μια έκθεση πρωτοβουλία και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ζήτησε την έκθεση ε, η έκθεση αξίζει δύο βαθμούς. Υπάρχει και μια επιστολή του Προέδρου της διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών που μας ζητούν ε, να ερμηνεύσουμε τα άρθρα 27 και 28 του κανονισμού. Οι συντονιστές προτείνουν να αποαντήσει ο πρόεδρος, να κάνει ο πρόεδρος την αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση είναι αρκετά απλή. Το ίδιο προτείνεται και σε ό,τι αφορά την επαλήθευση των προσωρινών μέτρων που αποφασίστηκαν τη διάσκεψη των Προέδρων τον περασμένο Μάιο. Επίσης, στην Επιτροπή μας ε, θέλουμε να συμμετάσχουμε μια αντιπροσωπεία στην ακρόαση του, του μελλοντικού αντιπρόεδρου της Κομισιόν υπεύθυνο για τις εξωτερικές υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των αρμοδιοτήτων του. Θα θέλαμε λοιπόν να είμαστε, να παρόντες σε αυτή την ακρόαση. Επίσης, συζητήθηκε αν θα χρησιμοποιήσουμε κονδύλια της Επιτροπής μας, είναι δυνατό αυτό, για μια έρευνα, ε, μια συγκριτική έρευνα για τα εκλογικά συστήματα των Ομοσπονδιακών κρατών. Όπως θα θυμάστε, μία από τις επιφυλάξεις που αναφέρεται από το συνταγματικό γερμανικό δικαστήριο σε ένα σημείωμα της 30 Ιουνίου είναι η απουσία ενός δημοκρατικού καθεστώτος ε, της, δημοκρατικής, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να δούμε τι συμβαίνει στα επιμέρους κράτη. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά στα ομοσπονδιακά κράτη, ε, για να δούμε ποια είναι τα εκλογικά του συστήματα. Μια και δεν υπάρχει ένα σύστημα δημοκρατικό, ένα ενιαίο δηλαδή σύστημα. Σε ό,τι αφορά την ε, προσχώρηση στη Σύμβαση για τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες, προτείνουμε να κάνουμε μια ακρόαση ε, που θα αποφασίσουμε ότι θα γίνει εν χρόνο. Θα γίνει μια επίσκεψη μια αποστολή μα στην Ουγγαρία το δεύτερο εξάμεινο του 2010 εν ώψη τη Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου. Και τέλο, προτείνεται να οργανώσουμε διάφορε επισκέψει αντιπροσωπιών τη Επιτροπή μα σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα, μέσα στην επόμενη πενταετία. Θα ξεκινήσουμε από κάποιες χώρες την επόμενη χρονιά, το 2010, και θα, θα συζητήσουμε το θέμα του μέλλοντος της Ευρώπης στις χώρες αυτές. Θα μιλήσουμε για την δημοκρατία, την ε, κυριαρχία και την εθνική ταυτότητα. Προτείνουμε την επόμενη χρονιά να πάμε στον Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πολωνία, στην Ιταλία και στη Γερμανία. Φυσικά όλες αυτές οι προτάσεις μπορούν να αλλάξουν μετά από τις παρεμβάσεις σας. Εγώ σας λέω ότι αποφασίστηκε στη μακρά συνεδρίαση τη χθεσινοβραδινή των συντονιστών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές είναι αποδεκτές, εγκρίθηκαν. Πολύ ωραία. Η Επιτροπή λοιπόν ε, συμφωνεί με τις προτάσεις των συντονιστών. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο για την ακρόση του Επιτρόπου υπεύθυνου για θεσμικές υποθέσεις. Στις 19 Οκτωβρίου είχαμε αρχίσει να συζητάμε, διορίζοντας τον συνάδελφο Τρασκόρση και για, για την ακρόαση εδώ και τον ε, κύριο Νταφ για το σύνολο των διαδικασιών ακροάσεων. Υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα ότι 25 Νοεμβρίου, 4 ε, Δεκεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ ταχείς. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα ότι η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προτείνει να υπάρχει ένα εκτιματολόγιο για όλες τις Επιτροπές ε, με μια εξαίρεση μπορούμε δηλαδή να προσθέσουμε ή να αντικαταστήσουμε κάποιες ερωτήσεις με πιο ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις που να σχετίζονται με τις προτεραιότητες της εκάστοτε ακρόασης, του εκάστοτε επιτρόπου. Έχετε το σχέδιο του ερωτηματολογίου, το οποίο ε, πονήθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων και με βάση αυτό μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Νομίζω ότι... Θα ήθελα ο Αντιπρόεδρος κ. Τσασκόφσκι να παρέμβει παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, για να μην επαναλάβω τα όσα είπε ο Πρόεδρος, θα σημειώσω ότι έχουμε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Μας ενημερώσαν άλλωστε ότι την ε, συζήτηση αυτή έπρεπε να την ετοιμάσουμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα που λείπαμε εκεί περισσότεροι και έτσι δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουμε τη συζήτηση. Κατά την ε, προετοιμασία λοιπόν αυτών των πέντε προτεραιοτήτων, μόνο μερικού από εσά μπόρεσα να βρω να επικοινωνήσω. Ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα και να προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες μας από κοινού. Για να επανέλθω στο ζήτημα μια μεταρρύθμιση που είχε προετοιμάσει ο, πρόταση για μεταρρύθμιση που είχε προετοιμάσει ο Αντζουντάφ από την προηγούμενη θητεία ε, και τις ε, ερωτήσεις για τους πέντε υποψήφιους επιτρόπους που είχαν προετοιμάσει οι επιτροπές. Όπως είπε και ο Πρόεδρος τώρα, είχαμε μια ολόκληρη συζήτηση για τη χρήση ενός ενιαίου ερωτηματολογίου με αρκετές διαφωνίες, κάποιοι είχαν αντιρρήσεις, αλλά και για λόγους των χρονικών περιορισμών όρισε η διάσκεψη των Προέδρων ότι θα ετοιμαστεί ένα ερωτηματολόγιο με πέντε ερωτήσεις που θα είναι ίδιες για όλους τους υποψήφιους επιτρόπους. Τις έχετε στο φακελό σας, είναι αρκετά γενικόλογη η διατύπωσή τους. Η πρώτη έχει να κάνει με το βιογραφικό του ίδιου του επιτρόπου, τις, ε, ε, τα προσόντα του κτλ η δεύτερη αφορά περισσότερο εμά, δηλαδή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου, όπω και οι υπόλοιπε. Και γενικά είναι ανοιχτά, ανοιχτή, αρκετά εμ, γενικόλογη διατύπωση, έτσι ώστε να μπορέσει ο κάθε επίτροπο να διατυπώσει τι δικέ του προτεραιότητε. Ε, δεν ήμασταν όλοι βέβαια ικανοποιημένοι με αυτή τη λύση και έτσι βρήκαμε το τη χρυσή τομή, λέγοντα ότι η κάθε επιτροπή θα μπορούσε συμπληρωματικά να προσδιορίσει ένα παράρτημα στην πέμπτη ερώτηση με τις δικές της προτεραιότητες και ερωτήσεις. Αυτό λοιπόν θα το κρίνουμε εμεί τώρα, αν θέλουμε να διατυπώσουμε συστάσει ή αν θέλουμε να προσδιορίσουμε προτεραιότητε. Εγώ προτείνω προτεραιότητε. Αλλά φυσικά αυτό το συζητάμε. Θα ήταν μάλλον δύσκολο να προσδιοριστούν ε, ε, συστάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στη δική μας περίπτωση, αλλά αυτά τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά, αλλά μπορούμε να το συστήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτιμώ προτεραιότητες για την πέμπτη ερώτηση. Χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, ε, είναι αρκετά στενά τα όρια τα χρονικά. Μέχρι το τέλος της, επόμενης, της ε, εβδομάδας πρέπει να είμαστε έτοιμοι. όπω είπε και ο πρόεδρο πρέπει να εργαστούμε πολύ γρήγορα. Και από την άλλη έχουμε δυσκολία και προ τι ίδιε τι ακροάσει, αλλά θα μα διαφωτίσει μάλλον ο Άντριου πιο διεξοδικά. γιατί φαίνεται ότι θα είναι μάλλον αδύνατον να ολοκληρωθεί η διαδικασία όλων των ακροάσεων μέσα στο Δεκέμβριο. Ίσως χρειαστεί να τις παρατείνουμε μέχρι και τον Ιανουάριο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχετε δει τις ερωτήσεις που έχουν, προτείνει, που έχουν προταθεί για το ερωτηματολόγιο. Αν θέλετε να τις δούμε μία-μία και πάλι με την επισήμανση ότι αρκετός χρόνος για συζήτηση και προετοιμασία δεν δόθηκε και άρα εγώ κάνω μία πρόταση αν θέλετε για να συμβάλλω στη συζήτηση και ασφαλώς ε, μπορείτε να κάνετε αντιπροτάσεις και τροποποιήσεις έτσι ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αλλά επαναλαμβάνω για τρίτη και ελπίζω τελευταία φορά ότι αρκετό χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, προτεραιότητες πρώτη προτεραιότητα παρακολούθηση των, της θέσης Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, κοινοβουλευτική εξέταση της, εξωτερικής, ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, όπως ορίζεται στην έκθεση για τις θεματικές πτυχές ε, της θέσπισης της σχετικής υπηρεσίας. Δεύτερον, εφαρμογή νέων στοιχείων που εισάγονται με την συνθήκη της Λισαβόνας σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια εν ώψη του νέου μηχανισμού ενισχυμένου ελέγχου με την αρχή της επικουρικότητα τη τάση της επικουρικής χρήση, τη λεγόμενη κίτρινη κάρτα, το λεγόμενο νέο σύστημα χειρόφρενου ή κατεπίγους ε, στροχοπέδησης και το σύστημα της ε, επιτροπολογίας. Το Βουλίες Πολιτών, Ρήτρα, ε, Έχουμε επίση την εφαρμογή του προγράμματο τη Στοκχόλμη, έχουμε επίση το σύστημα, την επανεξέταση μάλλον του εκλογικού δικαίου και στην υπαριθμόν 5 ερώτηση την άσκηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Εξουσιών του για ε, διατύπωση αιτήματο ε, νομοθετική πράξη από την Επιτροπή από το, το νέο άρθρο 225. Άρα εδώ έχουμε προσθέσει εξουσίε σε πρακτικό επίπεδο. Αυτές είναι οι πέντε προτάσεις. Αν θέλετε μπορούμε να τις συζητήσουμε. φυσικά πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Πρώτα απ' όλα, αν θα περιοριστούμε σε ε, συστάσεις, αν θα ε, περιοριστούμε σε προτεραιότητε, αν θέλουμε να είμαστε πιο γενικόλογοι ή πιο συγκεκριμένοι. Υπαγραμμίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητες ή συστάσεις, όπως μας είπε η Επιτροπή των ε, η διάσκεψη των Προέδρων, μπορούμε να είμαστε κάποιοι συγκεκριμένοι σε κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά βέβαια έχουμε και το θέμα του περιεχομένου τη ουσία, δηλαδή ε, στη συνέχεια να δούμε εφόσον καταλήξουμε ότι θέλουμε προτεραιότητες πρέπει να δούμε αν συμφωνούμε με το περιεχόμενο τους αν αυτές είναι πράγματι οι πιο σημαντικές, οι πιο σημαντικοί τομείς και εάν είναι οι πιο σημαντικοί τομείς τη σειρά με την οποία θα τους απαριθμίσουμε γιατί μπορεί μια ερώτηση να έρθει πιο μπροστά από την άλλη να θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντική κτλ. Αυτά. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας ε, για να καταλήξουμε στι ερωτήσεις που θέλουμε να υποβάλουμε στον Επίτροπο. Πριν ξεκινήσετε όμως, ίσως θα ήταν καλό να δούμε λίγο τις γενικές, την πρώτη κατηγορία ερωτήσεων, τις πέντε γενικές ε, κατηγορίες ε, ερωτήσεις, γιατί οι παριθμό 4 και 5 αναφέρονται στις απόψεις του υποψήφιου ε, ως προς τις προτεραιότητες ε, και οι δύο και τρία ως προς τις ε, σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο κύριος Ντάβ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ως προς το χρονοδιάγραμμα. Η διαδικασία προβλέπει ότι όλοι οι διορισμοί, το πακέτο των διορισμών θα εγκριθεί σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αν όχι στις 12 του μηνός, ίσως και λίγο νωρίτερα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος Μπαρόζο θα ζητήσει κάποιο χρόνο για να κατανείμει τις αρμοδιότητες ε, στους επιτρόπους, τα χαρτοφυλάκια τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Μακάρι να γινόταν γρήγορα, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο θα φανταζόμαστε να γίνει η κατανομή των χαρτοφυλακίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει τα ερωτηματολόγια του μετά την πρόταση που θα υποβάλει ο πρόεδρος Μπαρόζο για, την, για τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων. Μετά την αποστολή των ερωτηματολογίων, οι υποψήφοι επίτροποι δικαιούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγια του Κοινοβουλίου. Και φυσικά για να ενημερωθούν για το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Και ίσως ε, ορισμένοι υποψήφοι επίτροποι θα ενημερωθούν ε, πιο γρήγορα και θα, ενημερω... θα ετοιμάσουν πιο γρήγορα τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, αλλά αν θέλουμε να σεβαστούμε τη σοβαρότητα της διαδικασίας αυτής και την αξιοπιστία των ακροάσεων, θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε μια προσεκτική προετοιμασία και από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διεξαχθούν εύρυθμα και οι ακροάσεις. Οι απαντήσεις άλλωστε στα ερωτηματολόγια θα πρέπει να μεταφραστούν σε πολλές γλώσσες, κάτι που θα παρατείνει τη διαδικασία. Οπότε οι ακροάσεις δεν μπορούν να αρχίσουν πριν ε, την ε, Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Και σίγουρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό και θα πρέπει να προγραμματίσουμε την ολοκλήρωση των ακροάσεων στις αρχές του Ιανουαρίου, το αργότερο. Αν θέλουμε η επίσημη έγκριση του Συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να γίνει με βάση το πρόγραμμα. Και άρα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. και παρόλο που μπορούν να, να διεξαχθούν εκ παραλλήλου δύο ακροάσεις, δεν είναι προτιμότερο κάτι τέτοιο. Γιατί και το Κοινοβούλιο και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις ακροάσεις και των 26 υποψηφίων. Και αν συμπίπτουν οι ακροάσεις θα είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. και η διεξαγωγή παράλληλων ακροάσεων παρακολεί τη δυνατότητα παρακολεί δυνατότητα διεξαγωγής εξονυχιστικού ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτεραιότητες της Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που μας πρότεινε ο εισηγητής Ράφαου Τσασκόφσκι. Παραλείπεται ένα τμήμα που αφορά την ευθύνη του αρμόδιου επιτρόπου για τις ε, διοργανικές σχέσεις και τις ε, εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού. Η Επίτροπος Βάλστρομ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες και τα έγγραφα της Ένωσης. και προσπάθησε να ενισχύσει τη συνεργασία Συμβουλίου, ε, Κοινοβουλίου συγγνώμη, και Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, να βελτιωθεί η διαφάνεια και η εντύπωση που έχουν οι πολίτες για την Ένωση. Οπότε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια ερώτηση για το ποια είναι η γνώμη του υποψήφιου επιτρόπου σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, την καλύτερη πρόσβαση και ενημέρωση του κοινού για τα κοινοτικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την ε, εκλογική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, αυτό το σημείο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Αλλά ας μην είμαστε ιδιαίτερα κατηγορηματικοί στο στάδιο αυτό. Γιατί μια τέτοια μεταρρύθμιση προϋποθέτει εκτενείς διαβουλεύσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με τα εθνικά κοινοβούλια, με τα πολιτικά κόμματα. Και από τις διαβουλεύσεις αυτές θα διαπιστώσουμε αν υπάρχει έδαφος για συνένεση σε τόσο ευαίσθητα θέματα. και μία ερώτηση για το τι σημασία τι θα δώσει ο Επίτροπος, ο υποψήφιος Επίτροπος σε θέματα της μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος. Μια γενική ερώτηση όμως για το θέμα αυτό είναι σημαντική. Αλλά να είναι σχετικά ε, γενική και αφηρημένη και όχι πολύ συγκεκριμένη γιατί τι είδους μεταρρυθμίσεις συγκεκριμένα περιμένουμε από τον Επίτροπο. Αλλά μια τέτοια ερώτηση γενικά διατυπωμένη χρειάζεται. Κατά του λοιπού συμφωνώ με τον κατάλογο των προτεραιοτήτων της Επιτροπής μας, αν και πιστεύω ότι το σημείο 5 θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την ερώτηση για το πρόβλημα κακής ενημέρωσης των πολιτών, η βελτίωση της επικοινωνίας και της διαφάνειας με τους πολίτες. Πριν δώσω το, το λόγο στο συνάδελφο κ. Γιώργο Στέγκουι, θα ήθελα να θέσω επιτάπητο όλα τα στοιχεία της συζήτησης. Όλες οι συζητήσεις μας και τα αποτελέσματα των συζητήσεων μας θα, θα ανακοινωθούν μέχρι τις 6. Οι υπηρεσίες μας μας ανακοινώνουν ότι η διάσκεψη των Προέδρων θα μπορούσε να θέσει αυτό το ενιαίο ερωτηματολόγιο στη διάθεση των ε, υποψηφίων επιτρόπων τη στιγμή που θα συγκληθεί το Σώμα των Επιτρόπων ή και πριν, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι για τη βδομάδα 30 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου. Αυτά μας λένε οι υπηρεσίες μας. Ο κύριος Δεν μπορώ να λέει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τσασκόφσκι που μας ε, υπέβαλε μία πλήρη δέσμη ερωτήσεων που θα αποτελέσουν χρήσιμη βάση για την ε, εξέταση της καταλληλότητας του Επιτρόπου. Έχω όμως μία αμφιβολία. Όταν θα έρθει ο Επίτροπος, ο υποψήφιος Επίτροπος στην, Επιτροπή Τι θα εξετάσουμε, την καταλληλότητά του ή το πρόγραμμα της κυβέρνησής του. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ακολουθώντας α, τη σύσταση σύνεσης που μας έκανε ο συνάδελφος Νταφ, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στόχος της εξέτασής μας είναι όχι το οι προγραμματικέ δηλώσει του Επιτρόπου, αλλά η καταλληλότητα για την ανάληψη των ευθυνών του. Δεν μας ενδιαφέρει να μας δώσει απάντηση για όλα τα πολιτικά προβλήματα που απασχολούν την Επιτροπή μας, αλλά το κατά πόσο είναι κατάλληλο για αυτή τη θέση. Προσοχή λοιπόν και φρόνηση ως προς τις ερωτήσεις, για να δούμε και τι διατύπωση θα υιοθετήσουμε. Και μια άλλη παρατήρηση για τις ερωτήσεις. Από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί, θα γνωστοποιηθεί ο υποψήφιος για τα θεσμικά θέματα, θα συγκεκριμενοποιηθούν και πολλά θέματα καταλληλότητας. Η εθνική του θέση, η πολιτική του στάση απέναντι σε ορισμένα πολιτικά ζητήματα, το ιστορικό του, το βιογραφικό του από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση για το ποιος είναι υποψήφιος, ε, θα δούμε με βάση τις γνώσεις που θα συλλέξουμε για το πρόσωπό του, πώς θα διαμορφώσουμε και τις ερωτήσεις. Γιατί άλλο να έχουμε υποψήφιο από μια ευρωσκεπτιστική χώρα και άλλο να έχουμε υποψήφιο από μια φεντεραλιστική χώρα ή χώρα που είναι υπέρ της ε, φεντεραλιστικής δομής της Ένωσης. Είναι σημαντικό να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά. Για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα έχω κάποια σχόλια. θα πρέπει από τον υποψήφιο την υποψήφια επίτροπο να θέσουμε μια ερώτηση για να δούμε κατά πόσο είναι κατάλληλος αυτός ο υποψήφιος να ασκήσει το αξίωμα του Επιτρόπου ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιρροές της χώρας του. Θα πρέπει να περιμένουμε από έναν Επίτροπο να αναλάβει έναν ευρωπαϊκό ρόλο πρώτα απ' όλα. Να απομακρυνθεί από τους όρους και τις πολιτικές συνθήκες της χώρας που τον διόρισε. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει έναν γνήσιο ευρωπαϊκό ρόλο. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν οι επίτροποι από τα εθνικά τους συμφέροντα από τα συμφέροντα της χώρας τους και αυτό είναι βασικό στοιχείο για να ελέγξουμε την καταλληλότητά τους για τη θέση αυτή. Μία ερώτηση που μας βασανίζει χρόνια ολόκληρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σχέση του Επιτρόπου, η θέση του Επιτρόπου απέναντι στην εξίσωση Ευρώπη πολίτης. Αυτή η εξίσωση είναι πολύ σημαντική. Αυτή η σχέση είναι πολύ σημαντική γιατί όλοι έχουμε επίγνωση του αβυσαλαίου χάσματος που χωρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τεράστια απόσταση της Ένωσης από τον πολίτη. Και για να καλύψουμε, να γεφυρώσουμε αυτό το κενό, χρειαζόμαστε μια πολιτική. Ίσως αυτή η ερώτηση θα μπορούσε να τεθεί στον Επίτροπο. Πώς σκοπεύει να γεφυρώσει αυτό το κενό. Έχουμε και μια άλλη σημαντική εξίσωση οικονομική κρίση και πολιτική κρίση και οι σχέσεις τους με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Γιατί δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε μπροστά στην πραγματικότητα αυτή. Η οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση και η συμπερίληψη της πολιτικής σε διάφορους τομείς οδηγεί τη σχέση, οδηγεί σε διέξοδο τη σχέση του πολίτη με την πολιτική και του πολίτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή μας και υπό αυτό το πρίσμα να ελέγξουμε την και υπό αυτό το πρίσμα να ελέγξουμε την καταλληλότητα του Επιτρόπου. Τέλος, θα πρέπει να εξετάσουμε και κάτι που ίσως δεν είναι το χειρότερο κακό, αλλά αναφέρθηκε χθε ω παράπονο ότι πρόκειται για τη δυνατότητα αυτοεξαίρεση τριών χωρών από, την, από το Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Οι τρει αυτές χώρες είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Πολωνία και η Τσεχία. Όταν προσχωρήσει η Κροατία και θα πρέπει να εγκρίνει το πρωτόκολλο ένταξης τη Τσεχίας ή μέχρι τότε μπορούν και άλλε αυτοεξαιρέσει να προταθούν. Ποια είναι η θέση του Επιτρόπου απέναντι σε αυτή την, κατά τη γνώμη μου, αξιοθρύνητη στάση της αυτοεξαίρεσης ορισμένων χωρών από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ας μην ξεχνούμε και την απόφαση του Συνταγματικού Γερμανικού Δικαστήριου. Έχουμε πει πολλές φορές στην Επιτροπή μας ότι μία από τις νομικές βάσεις της ε, απόφασης αυτής δημιουργεί επικίνδυνη αφισβήτηση των θεμελίων της Ένωσης και της ίδιας της νομιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον Επίτροπο πώς τοποθετείται απέναντι στο θέμα αυτό, την απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου και ποιες είναι οι προβλέψεις του, οι προθέσεις του για να αντιμετωπίσει τέτοιες βαθιά αντιευρωπαϊκές τάσεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα θίξουμε στην ακρόαση με τον υποψήφιο επίτροπο. Τώρα μου ζήτησε το λόγο για μία στιγμή να παρέμβει ο εισηγητής Τσασκόφσκι να θέσει κάποια στοιχεία διακόπτοντας τη ροή των παρεμβάσεων, των κανονικών παρεμβάσεων, αλλά για μία στιγμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλησα να μακρηγορήσω στην εισαγωγική μου παρέμβαση, αλλά ίσω χρειάζεται να πούμε μερικά λόγια ακόμα ως προς την ε, κατάσταση που έχουμε μπροστά μας, για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε λίγο στη συζήτηση. Πρώτον, και πιο σημαντικό, έχουμε να κάνουμε με γραπτές ερωτήσεις. Συζητούμε τι γραπτές ερωτήσει και πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι θέλουμε να επιτύχουμε με τι γραπτέ ερωτήσει. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια τη ακρόαση, διατυπώνουμε οποιαδήποτε ερώτηση θέλουμε για συγκεκριμένε πτυχέ όπω αυτέ που αναφέρατε. Επομένω, η αδίποτε πτυχή θεωρούμε σημαντική. Η ερώτηση σα φέρει γιατί ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, το μέλλον ε, σχετικά με το θέμα αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, θα μπορούσε να υποβληθεί ω προφορική ερώτηση, όπω και πολλέ άλλε. Άρα αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε τις πέντε δικέ μας προτεραιότητες ε, σε σχέση με τον ε, ή την Επίτροπο. Άρα, Περισσότερο μιλούμε για πιο γενικέ ερωτήσει Πολύ ευχαριστώ να αλλάξουμε αν θέλετε κάποια διατύπωση, να τροποποιήσουμε, αλλά βάλουμε άλλη ερώτηση αντί για αυτέ που έχουμε συμπεριλάβει στον κατάλογο. Αλλά δεν μπορούμε να συζητούμε ε, έναν ατέρμονο κατάλογο προφορικών ερωτήσεων, γιατί αυτές θα τις δούμε στην προφορική ακρόαση. ακρόαση. Κατά τα άλλα, θα ήθελα και θα σας το διαβάσω ε, ή τουλάχιστον σας περιγράψω το περιεχόμενό τους να σας αναφέρω τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτέ οι γενικόλογε ερωτήσει που έχει προσδορίσει στις διάσκεψη των Προέδρων και σα τα διαβάζω. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση, η οποία υποβάλλεται σε όλου του ε, επιτρόπους ε, υπογραμμίζω, έχουν να κάνουν με την προσωπική ανεξαρτησία και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ένας επίτροπος. Δηλαδή, τι είδους, ε, από, τα, ποια από τα δικά σα προσόντα μπορούν να σα βοηθήσουν στη δουλειά στους επιτρόπου να προαγάγετε το κοινό κοινοτικό συμφέρον, τι είδου εχέγγυα ανεξαρτησία σα θα να παρουσιάσετε και ούτω καθεξή. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε εσεί προσόντα ανεξαρτησία εργασία, στην, ε, στη δουλειά και όλα αυτά είναι μέσα στο γενικό ερωτηματολόγιο τη δέσκευση των Προέδρων. Οι άλλε δύο ερωτήσει έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι επιτροπέ αυτού. Ε, παραδείγματι, πώ αξιολογείτε το ρόλο σα ω ε, μέλο του συλλογικού οργάνου ε, τη Επιτροπή και πώ θεωρείτε ότι είσαστε υπόλογο έναντι του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν μέσα στην κατάλογο. Τι είδου δεσμεύσει μπορείτε συγκεκριμένα να λάβετε ω προ την ενίσχυση τη αδιαφάνεια, τη συνεργασία και ούτω καθεξής και σε ποιο βαθμό μπορείτε να προσφέρετε, να δεσμευτείτε ότι θα προσφέρετε τις ε, απαραίτητε πληροφορίες και έγγραφα στις διαδικασίες στο Κοινοβούλιο. Και επίσης συνεχίζω πώς μπορείτε να υλοποιήσετε τα καθήκοντά σα μέσα από το χαρτοφυλάκι που σας έχει ανατεθεί. Αυτά λοιπόν είναι οι γενικές ερωτήσεις για να παρουσιάσει ο κάθε ένας ε, επίτροπος τα χαρακτηριστικά του, το χαρακτήρα του, τις ικανότητές του. Όπως είπατε και εσείς κύριε Γιάρεγγι, είναι ο κάθε άνθρωπος διαφορετικός, έχει διαφορετική προσωπικότητα και χαρακτήρα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να δούμε πώς βλέπει το ρόλο του, πώς βλέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς βλέπει τις διοργανικές σχέσεις. Και στη συνέχεια ε, θα μπορέσουμε ασφαλώς ε, να τον χόρεψουμε στο ταξιψί με τις προφορικές μας ερωτήσεις ε, για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Γενικές ερωτήσεις λοιπόν τις έχουμε, έχουμε καλύψει τα θέματα. Στις πιο ιδιαίτερες ερωτήσεις, πιο ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούμε μέσα από την προφορική διαδικασία να τις καλύψουμε. Εγώ αυτό που θέλω είναι να προσδορίσουμε τις πέντε για μας πιο σημαντικές προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να δώσει απαντήσει ο Επίτροπος. Και μια και δεν έχουμε χρόνο, ας επικεντρωθούμε σε αυτά για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε μια κοινή θέση, τις πέντε αυτές ερωτήσεις μας, να τις αναδιατυπώσω, να σας τις υποβάλω και πάλι και έτσι άτυπα έστω να προσπαθήσουμε να τις επεξεργαστούμε σήμερα αύριο, να είμαστε έτοιμοι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο και εισηγητή κύριο Τσασκόφσκι για την ε, σαφήνειά του, γιατί κάνει αυτή τη διάκριση ανάμεσα στις γενικές ερωτήσεις και στις ειδικέ ερωτήσεις που θα είναι προφορικές. Και οι προτεραιότητες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο, όπως αναφέρει και το ερωτηματολόγιο, ιδίω τα πολιτικά θέματα. Αναφέρονται λοιπόν στο ενιαίο ερωτηματολόγιο. Ο Σέπλινγκ ζητάει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Τσασκόφσκι για την δουλειά που έκανε και για τη διευκρίνηση που μόλις μας έδωσε. Ε, νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα γενικά ερωτήματα και στα ερωτήματα τα οποία φτιάξετε εσείς για να τα εξετάσει η Επιτροπή μας. Η Επιτροπή μας. Είναι η σχέση μεταξύ των δύο που με ανησυχεί λιγάκι και θα ήθελα να τη σχολιάσω. Καταρχάς, ε, στις ερωτήσεις σας δεν υπάρχει τίποτα για αυτό που θεωρώ θεμελιώδη διάσταση της δουλειάς της Επιτροπής μας. Δηλαδή, το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχει μέσος, αλλά όχι ε, σαφώς. Α, αξίζει να το καταστήσουμε σαφές. Γιατί για μας, για την ακρόαση, θα κάνουμε ερωτήσεις πώς ο υποψήφιος επίτροπος ε, προσδιορίζει το ευρωπαϊκό συμφέρον και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Κατανοεί την εργασία που κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό θέτει ερωτήματα σχέσεων με τους πολίτες βεβαίως. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι σωστό να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, και αυτό θα το κάνουμε όταν ξέρουμε τα ονόματα, το ιστορικό του ε, επιτρόπου στη χώρα του, η χώρα της. Γιατί αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο που θεωρούμε αυτό το άτομο και είναι πολύ πιθανό α, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κατανοεί το πλαίσιο της εντολής που θα λάβει. Μια άλλη ερώτηση αφορά τις προτεραιότητες. Ε, είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν τρεις. Ε, σωστό, υπάρχουν και στην βασική επιστολή. Αλλά αυτές που αναφέρατε, πώς θα τις συντονίσουμε, δηλαδή πώς θα τις ιεραρχήσουμε. Ε, μέσα σε τι χρονοδιάγραμμα, από ποιων πολιτικών, γιατί επηρεάζεται η μία από την άλλη. Ε, υπάρχει σχέση αιτίου, του. Αν ξεκινήσει με τη μία, ας πούμε, πώς προωθείται η άλλη κτλ. κτλ. Τέτοιου τύπου ερωτήσεις, δηλαδή. Πρόεδρος. Ο κύριος Μακμίλαν Σκότ, ο αντιπρόεδρο, έφτασε. Δεν έχει όμω πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Έχει και άλλα καθήκοντα. Αν λοιπόν συμφωνείτε να σταματήσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση που διεξάγουμε τώρα για το θέμα των ακροάσεων των επιτρόπων και ιδίω του αρμοδίου επιτρόπου που θα ασχοληθεί με θέμα της Επιτροπής μας και να περάσουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα επανέλθουμε στην ερώτησή στο, στη συζήτησή μας όταν φύγει ο αντιπρόεδρος ε, Μακμίλαν Σκότ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το σημείο 5. Όπως θα ξέρετε, η ΚΟΖΑΚ συνεδρίασε στη Στοκχόλμη το Σεπτέμβρη, α, όχι λάθος, 5 με 8 Οκτωβρίου, λέει ο Πρόεδρος. Και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είχε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο ακριβώς Μακμίλαν Σκότ. Ε, μοιράστηκαν οι φάκελοι για αυτή την συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ. Ε, φαντάζομαι έχετε τα σχετικά κείμενα στα αγγλικά και στα γαλλικά και το κείμενο των παρεμβάσεων και το κείμενο των συμπερασμάτων. Θα ήθελα ο Αντιπρόεδρος λοιπόν να μας παρουσιάσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ε, είναι ιδιαίτερη τιμή που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα για την τελευταία συνεργασία της ΚΟΖΑΚ. Ξέρετε ότι ήταν παρόν ο πρόεδρό σα επίση στη σε αυτή 4, και 4 με 6 Οκτωβρίου στο Εκχόλμη. Η ίδια η συνεδρίαση είχε μέλη ε, εκπροσώπους και των Εθνικών Κοινοβουλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές και, τον και της Άνω και της Κατοβουλής και έλεγε χώρα μέσω σχεδόν μετά τα, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ιρλανδικού ε, δημοψηφίσματος και ασφαλώς ε, αυτό έγινε δεκτό με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τους συνέδρους. Τώρα έχουμε δύο αντιπρόεδρους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολούνται με τα θέματα αυτά που καθοδηγούν την πορεία αυτή. Εγώ είχα την τιμή και, στις δύο, και στην τελευταία θητεία να έχω αυτή την ε, θέση. Λόγω της συνεδρίασης του Προεδρίου ταυτόχρονα στο Παρίσι, στον Νίκο Ζαμονέ, δεν ήταν ε, ο άλλος αντιπρόεδρος ε, στην ε, Κόζα εγώ όμως ήμουν παρόν, όπως άλλωστε έχω παρακολουθήσει όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων για μένα έχουν τεράστια σημασία. Όπως γνωρίζει η Επιτροπή σας, γίνονται συζητήσεις για την εκπροσώπηση στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδριάση της ΚΟΖΑΚ. Εγώ ε, μπορώ ευχαριστώ να συστήσω κάθε επιλογή. Η Επιτροπή σας μπορεί να καθοδηγήσει τις, ε, τους χειρισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα που ε, υπάγονται στην Λισαβόνα. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης λύσης, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω το Κοινοβούλιο βρίσκεται στη μοναδική πλειονεκτική θέση ως προς το ότι είναι το μόνο μόνιμο μέλος της Τρόικα τη Κόζακ και παράλληλα επιτρέπει και τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την ε, γραμματεία της ε, Κόζακ, το γεγονό ότι είμαστε εδώ στι Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν, η συνεδρίαση έλαβε χώρα σε οικείο κλίμα, σε ευχάριστο κλίμα μετά την ανακοίνωση από τους Ιρλανδούς εκπροσώπους. Μετά ακούσαμε τον κύριο Ράινφελτ από τον, τον πρόεδρο, τον προεδρεύοντα της, ε, τη Σουηδία. Ακούστηκε η πρόβλεψη ότι θα επικυριωθεί το ταχύτερο δυνατό ε, η συνθήκη της Λισαβόνας και θα μπορέσουν να ληφθούν οι αποφάσεις από το Συμβούλιο ε, κορυφής για τα νέα πρόσωπα, για τους νέους θεσμούς που ιδρύονται. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε πρόταση για την ε, λεγόμενη συμβολή που είναι το επίσημο έγγραφο που ετοιμάζει η COSAC, Contribution, ως προς την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Προτείνουμε λοιπόν και έγινε δεκτό μια τροπολογία όπου λέμε δεδομένης της ε, έγκρισης συνθήκης Λισαβόνας από όλες τις βουλές των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, παρότι ακόμη ε, εκρεμεί το ζήτημα της ε, τυπικής κύρωσης από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο της συνθήκης ύστερα από την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος στις 2 Οκτωβρίου θεωρεί η Κόζακ ότι θα πρέπει να προχωρήσει εφόσον έχουν τηρηθεί οι θεσμικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την κύριο συνθήκη Λισαβόνας σε όλες τις χώρες μέλη, ε, το ταχύτερο δυνατό η συνθήκη. Αυτό ήταν μια έκκληση προς τους ε, ομόλογους μας της Πράγας όπως αντιλαμβάνεστε αλλά ευτυχώς εχθές ο πρόεδρος της ε, Πράγας ανεγνώρισε ο πρόεδρος της Τσεχίας ανεγνώρισε την ε, ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και τυπικά προχώρησε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και τυπικά και πρόεδρε θα ήθελα μια πολύ απλή πρόταση να υποβάλλω, μου επιτρέπετε. Οι λέξεις που απαρτίζουν τον τίτλο «Κόζακ» είναι λέξεις που έχουν επιλεγεί εδώ και πολύ καιρό, ναι, έχουν βαρύτητα, ναι, αλλά δεν γίνεται αντιληπτό ακριβώς το τι εκπροσωπεί η Κόζακ εύκολα. Και γι' αυτό εγώ θα πρότεινα να ε, αλλάξει το όνομα σχετικά σύντομα της ΚΟΖΑΚ, ίσως σε κοου-παρλ έτσι ώστε να φαίνεται ότι είμαστε ένα όργανο συνεργασίας κοινοβουλίων. Αλλάζει ο ρόλος της άλλωστε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε μια σχέση εταιρική και όχι ανταγωνιστική με τα εθνικά κοινοβούλια. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε απόλυτα την, ε, το νόμιμο έρισμα των Εθνικών Κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ, όπως ξέρετε, εκλέγομαι ως ανεξάρτητος πλέον, ε, αλλά συντηρητικός Βρετανός βουλευτής, ύστερα από διαφωνίες με το κόμμα μου, ε, είμαι άστεγος κομματικά, αλλά χάρη στη δική μου παρέμβαση και προσφυγή ανακοινώθηκε από, και από το κόμμα ότι αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας κυρώσεως και ως εκ τούτου παρετείται από, την, από το δημοψήφισμα, την πρόθεση δημοψηφίσματος. Ε, ωστόσο, ακούγονται κάποιες φωνές για μία άτυπη δημοσκόπηση ή άτυπη έγκριση από το λαό του ε, της συνθήκης, αν και ελπίζω ότι η ηγεσία του κόμματος μου, των συντηρητικών της Βρετανίας, θα αναγνωρίσει ότι πλέον χρειαζόμαστε την αναγνώριση της νομιμότητας, της, του νόμιμου έρασμου, ερίσματος ε, της συνθήκης Λισαβόνας. Είναι μια συνθήκη που από εωβαίνει όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει πλέον να τεθεί σε ισχύ και είναι η ώρα να τεθεί σε ισχύ τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση με παρεμβάσεις των συναδέλφων. Πρώτος ο κύριος Μπροκ. Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς τον συνάδελφο κύριο Αντιπρόεδρο. Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων και η ενίσχυση αρχή τη επικουρικότητα είναι ασφαλώ πολύ σημαντικά ζητήματα. Όπως άλλωστε και το ζήτημα της συνεργασίας στην παραγωγική διαδικασία εν γέννη. Τόσο στην διαδικασία παραγωγής των νομοθετημάτων, όσο και στην εκτέλεση αυτών σε επίπεδο κρατών μελών. Όλα θα κρυθούν από τη συνεργασία. Πλην όμω, δεν γνωρίζω εάν η COSAC είναι μακροπρόθεσμα ένα ε, εργαλείο πάνω στο οποίο μπορούμε να, συνεργαστούμε, να στηριχθούμε για τέτοιου είδου συνεργασία. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων. Η δε έννοια της συνεργασίας ως προς την αρχή της επικουρικότητας και την ε, υλοποίηση των ε, θεσμικών των νομοθετημάτων προϋποθέτει εμπλοκή και των ειδικευμένων μονάδων ή θεσμικών οργάνων των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν το να αλλάξει όνομα το κόπα, ε, η Κόζα Ξεκόπαρλ όπως προτείνει ο Αντιπρόεδρος ίσως να σημαίνει ότι θα μετατραπεί η Κόζα σε ένα είδος ε, διακοινοβουλευτικής διάσκεψης στην Ευρώπη πράγμα το οποίο εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερο γιατί σε αυτή την ε, σε αυτή την οργάνωση, σε αυτή τη δομή της ΚΟΖΑΚ είμαστε μόνο ένας από τους 28. Μόνο ένας από τους 28. Ενώ, δυνάμει της συνθήκης, είμαστε η πραγματική νομοθετική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ουσιαστική νομοθετική αρχή. Άρα λοιπόν το να εκχωρήσουμε εξουσίες και, ε, ε, ε, παρετούμενοι από, την, από τα δικαιώματα ή τις προνομίες μας ως νομοπαραγωγικού οργάνου και να γίνουμε μόνο το νούμερο ε, ε, μία μονάδα από τους 28 της ΚΟΖΑΚ νομίζω ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας. Και γι' αυτό θα πρότεινα η ΚΟΖΑΚ να μην λάβει ερμηνείες που ξεπερνούν τα όρια της συνθήκης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πρωτόκολλο της, ε, στη συνθήκη, ένα προσάρτημα στη συνθήκη και, και τίποτε περισσότερο. Και καλό θα ήταν να συζητήσουμε ήρεμα, αν θέλουμε, με χρόνο δηλαδή αρκετό, το πώ θέλουμε να προχωρήσει η ΚΟΖΑΚ. Επίση, οι αντιπρόεδροι, και ξέρει ότι δεν εννοώ εσένα προσωπικά, γιατί δεν, δεν είναι δυνατόν να εννοώ εσένα προσωπικά. Είναι, είναι σωστό το ότι εσύ είσαι ο αντιπρόεδρος που ασχολείται με τα θέματα αυτά αυτή την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, Ωστόσο όλα τα κοινοβούλια εκπροσωπούνται στην ΚΟΖΑΚ με πρόεδρους ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών. Γιατί λοιπόν εμείς αλλάζουμε το πρωτόκολλο και έχουμε διαφορετική μεταχείριση στο θέμα αυτό από ό,τι τα άλλα 27 κοινοβούλια. Γιατί να στείλουμε αντιπρόεδρο και όχι πρόεδρο επιτροπής. Αυτό άλλωστε σχετίζεται και με τα όσα είπα και στην αρχή. Ότι αισθάνομαι πως ε, τάση ή η συνδεση του Κοινοβουλίου κατά αυτόν τον τρόπο με την ε, ΚΟΖΑΚ ε, θα πρέπει να γίνει σε ισότιμους όρους και πάντως σε επίπεδο ίσως ε, Προέδρων Επιτροπών ή Προέδρου Επιτροπής. Ίσως ο κύριος Καζίνη μαζί με τον κύριο Μακμήραν Σκότ, τον Αντιπρόεδρο, θα, είχαν, θα ήταν σκόπιμο να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ώστε να μην χάσουμε κομμάτι από τις, τις εξουσίες, τα, τα προνόμια μας στην υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο κυρία Γκουρμάη. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κυρία Αντιπρόεδρε. Φυσικά μας ενδιαφέρουν τα ονόματα, αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο το καλό περιεχόμενο και η αγαστή συνεργασία. Και νομίζω ότι με απέραντο επαγγελματισμό ασχολείται σε υψηλό επίπεδο με τα θέματα αυτά και με πολύ έγκυρο τρόπο ο αρμόδιος αντιπρόεδρος. Χθες ε, στη διάρκεια της συνεδρίασης ακούσαμε ότι υπέγραψε και ο πρόεδρος Βάτσλαφ Κλάους και έτσι ήρθε και το τελευταίο εμπόδιο για την κύρωση της συνθήκης όλα τα εθνικά κοινοβούλια ήταν υπέρ της συνθήκης, ακόμη και σε χώρες ε, που ήταν πιο περίπλοκη διαδικασία κύριο και δεν περιοριζόταν στην κοινοβουλευτική έγκριση. Πάντως, ε, η νέα συνθήκη της Λισαβόνας θα ενισχύσει την ε, δημοκρατικότητα, αρκεί φυσικά να γίνει σεβαστή και αρχή της επικορικότητας, όπως είπε ο κύριος Μπρόκ. Βέβαια έχουμε και το γερμανικό παράδειγμα και πολλές φορές έχουμε τα εθνικά συμφέροντα, αλλά το σύστημα συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικού Κοινοβουλίου θα πρέπει να λειτουργεί το, συνταμό, να λειτουργεί το συνταμότερο δυνατό, όπως πρέπει να συμβεί και μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών εδώ και στι χώρε μέλη. Έχουμε Τρόικα, Ισπανία, Βέλγιο και Ουγγαρία. Αυτέ οι τρει χώρε τη Τρόικα θα πρέπει να πρωτοστατήσουν ε, υπέρ τη σύσφυξη αυτών των σχέσεων και στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας να προωθηθούν αυτές οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις. Άλλωστε θα συνεδριάσει η Κοζά στην Ουγγαρία. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι τρεις χώρες της ε, Τρόικας να δώσουμε ύψιστη προτεραιότητα στις θεσμικές εξελίξεις. Αν συμφωνείτε με όλα αυτά, μπορείτε να στηριχθείτε σε εμά να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Επίσης ε, θα έχουμε στενές σχέσεις και με τον εθνικό αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που πλήττουν άμεσα την Ουγγαρία, που είναι η μόνη χώρα της νέας ε, που συμμετέχει στην Τρόικα. Ε, έχουμε το πρόβλημα της περιοχής του Δούναβη και όπως και η Ισπανία έχουμε χτυπηθεί από μαζική μεταναστευτική ροή. Θα ήθελα πάντω να ευχαριστήσω τον κύριο Μακμίλαν Σκότ για όλες τις προσπάθειες που κάνει, όχι μόνο για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία, αλλά και για τα θέματα τη ισότητα των φύλων. Σα ευχαριστούμε κυρία Γκουρμάη. Ο κύριος Ράγκελ. Σα ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο Μακμίλαν Σκότ για τα αίσια αποτελέσματα που πέτυχε και για τις προσπάθειες που έκανε στην Κοζάκ προκειμένου να επιταχυνθεί η κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες αυτές ήταν σημαντικές. Γι' αυτό ας μην υποτιμούμε το ρόλο που διαδραμάτισε η Κοζάκ και η επίδραση που ασκήθηκε στους Τσέχους από την Κοζάκ που ίσως οδήγησαν ε, στη, στα τελικά θετικά αποτελέσματα και της τσεχικής κύρωσης. Σε ό,τι αφορά την Κοζάκ πάντως, πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως η δική μας Επιτροπή, να δώσουμε προτεραιότητα στις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό του κυρίου Μπροκ. Αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε πολλά εθνικά κοινοβούλια, η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων δεν εξετάζει ενδελεχώς τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και εκεί θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ένα παιδαγωγικό ρόλο και να ενημερώσει τα, τα εθνικά κοινοβούλια να γίνουμε φορείς πληροφόρησης προς τις Εθνικές Βουλές και ίσως μια ισχυρή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΟΖΑΚ έχει νόημα για να δείξει τη θέση του απέναντι στις υπόλοιπες βουλές. Παρακολούθησα πολύ στενά αυτό το θέμα από την αρχή και η αξιολόγηση που κάνουμε σήμερα για το έργο των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι σημαντική γιατί πολλές φορές τα Εθνικά Κοινοβούλια ασχολούνται κυρίως με τα εθνικά ζητήματα και δεν αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ούτε έχουν μια συνέχεια στην εξέταση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Και εκεί θα είναι σημαντικό το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προσπάθεια ενημέρωσης και διαμόρφωσης μιας ε, νοοτροπίας, μιας παιδείας ε, μεγαλύτερης εμπλοκής στα ευρωπαϊκά ζητήματα και μεγαλύτερο ενδιαφέροντος για τα ευρωπαϊκά πράγματα από πλευράς Εθνικών Κοινοβουλίων. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που από συνταγματική άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν απομονωμένα συντάγματα. Κάθε συνταγματικό πλαίσιο και κάθε κράτος επηρεάζεται και από τα ευρωπαϊκά συνταγματικά θέματα αλλά και από τα συνταγματικά πλαίσια των άλλων χωρών. Κοιτάξτε για παράδειγμα τι επίπτωση μπορεί να έχει η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τα συντάγματα άλλων χωρών. Υπάρχει στενή διακοινοβουλευτική και διασυνταγματική κατά κάποιο τρόπο σχέση μεταξύ μας. Και από αυτή την άποψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και το πλεονέκτημα, αλλά έχει και συμφέρον να αναβαθμίσει τη σχέση του με τα, με Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι οι καλύτεροι μας σύμμαχοι στην προσπάθεια άσκησης δημοκρατικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε πρώιμη φάση. Θα πρέπει από την αρχή να γίνει ο έλεγχος ε, του κυβερνητικού έργου. Γιατί οι αποφάσεις ε, το κυβερνήσεων μέσα στο Συμβούλιο μπορεί να διεξαχθεί σε πρώιμο στάδιο από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και αυτή την παιδεία της ε, αξιολόγησης θα πρέπει να την καλλιεργήσουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια ως ε, αντιπάλους. Ούτε θα πρέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια να αντιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, εχθρό τους ή ως ανταγωνιστή τους. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Μακμίλαν Σκότ ε, το πολύ σαν ένα τέταρτο θα πρέπει να φύγει. Γι' αυτό θα ήθελα όλοι οι παρεμβαίνοντες να σεβαστούν το χρονικό όριο των δύο λεπτών για να μπορέσει να απαντήσει ο Αντιπρόεδρος. Κύριος Μπρόντς. Thank you. Uh, Mr. Macmillan... Ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ είπε ότι η δημοκρατική νομιμότητα της, του προγράμματος επικύρωσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλλά το πρώην κόμμα του, το κόμμα των συντηρητικών, καθώς και το κυβερνό κόμμα, το κόμμα των εργατικών στη Βρετανία, ε, δεσμεύτηκαν το 2005 ότι θα κάνουν δημοψηφίσματα. Και από ό,τι ξέρω, παρότι βεβαίω δεν ήταν ε, υποψήφιος αυτήν την εκλογή, δεν πήρε τις αποστάσεις του. Πώς λοιπόν τώρα ε, μπορεί να, να αυτά τα δύο κόμματα ότι είναι δημοκρατικά ε, και νόμιμα. Ε, δημοκρατία σημαίνει εξουσία του λαού και όχι των κοινοβουλίων. Ο Βρετανικός λαός γίνεται όλο και πιο έξαλλος από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ολόκληρη πολιτική τάξη. Ευχαριστώ. Äh, ναι, νομίζω ότι αν ε, ρίξουμε μια ματιά και στην ημερησία μας διαταξή θα ήταν ε, ίσως σκόπιμο αντί να κοιτάμε προς τα πίσω και να ξανα... να επαναλαμβάνουμε παλιές ε, μάχες, να κοιτάξουμε προς τα μπρος και να δούμε εάν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ο κύριος Μακτήλαν Σκοτ και ο κύριος Μπρόκ νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρουσε ιδέες να προβάλλουν. Και εγώ θα ήθελα προς, όσον αφορά εμένα προσωπικά να πω ότι η σχέση μας, η μας προς τα εθνικά κοινοβούλια είναι όλο και σημαντικότερη και ίσως θα έπρεπε να, να διατυπώσουμε τον τρόπο σύστασης των αντιπροσωπιών Όσο δεν αφορά εμάς το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, εκφράζουμε, να εκπροσωπούμεθα σε επίπεδο ουσιαστικής δουλειάς, δηλαδή της δουλειάς που γίνεται στις επιτροπές και δει την Επιτροπή για τα θέματα στα, σταγματικά θέματα. Ίσως λοιπόν αντί να συνεχίσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στο παρελθόν, να δείξουμε μια διαφορετική ε, πρόταση ως προς τη σύνθεση των ε, αντιπροσωπιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σάπλιν. Σύντομα. Ε, το έφεσαν πολλοί συνάδελφοι αυτό το θέμα της ε, διαβίβασης των πληροφοριών και της ενημέρωσης. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς ούτω ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά θεσμικά όργανα, δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια, να έχουν επαφή. Ε, τώρα, μου ήρθε μία σκέψη α, που προέκυψε α, από αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος. Ε, η Ουγγαρία είναι, έχει την Προεδρία το πρώτο εξάμεινο του 2011. Θα μπορούσαμε να έχουμε ομαδικές ε, συνεδριάσεις υπό την αιγίδα των ΚΟΖΑΚ του α, της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, το τρίο της Προεδρίας, δηλαδή της Τρόικα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα, θα τα πάμε καλύτερο. Ο κύριος Τσασκόφσκι. I just want to uh, draw Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο μεταβαλλόμενο αυτό το οποίο μετά τη θέση ισχύ της νέας συνθήκης και μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Έχω την αίσθηση ότι όταν ιδρύθηκε η ΚΟΖΑΚ ήταν ε, ε, μία από τις ελάχιστες δυνατότητες που είχαμε για διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια. Και γι' αυτό χρειαζόταν τότε τώρα και θελήσαμε να εξασφαλίσουμε μία επιρροή των Εθνικών Κοινοβουλίων στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αλλά έκτοτε έχουν αλλάξει πάρα πολλά και συμφωνώ με τον Έλμαρ Μπροκ ότι θα πρέπει πια να ξανασκεφτούμε από την αρχή τη σχέση μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί οι σχέσεις μας έχουν σοβαρέψει. Καταρχήν με την ε, συντακτική συνέλευση. Για πρώτη φορά ενεπλάκησαν τα εθνικά κοινοβούλια στις ε, τροποποίησεις και τη μεταρρύθμιση συνθήκη. Έχουμε επίσης για πρώτη φορά με τη συνθήκη της Λισαβόνας τη διαδικασία της κίτρινη κάρτα. Εκεί θα αρχίσουμε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια για την εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας και, της, ε, και την, κυρίως την έμπρακτη εφαρμογή τη αρχή επικουρικότητας. Έχουμε και άλλε εξελίξει ε, καλούνται οι πρόεδροι των ε, Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων, των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων ε, των διαφόρων κοινοβουλίων προσκαλούνται στις συνεδριάσεις ε, για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε λοιπόν όλο και μεγαλύτερη ευάθυνση και πολλαπλασιασμό των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί δεν θα έχουμε μόνο συνέβρεση και συζήτηση. Γιατί στην αρχή οι της Κοζάκ ήταν περισσότερο θεωρητικές. Τώρα θα γίνουν πιο πρακτικές. Έχουμε πια νέες διάβλους επικοινωνίες και δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Και αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη μελλοντική μορφή της ΚΟΖΑΚ και τις μελλοντικές της λειτουργίες. Ευχαριστώ. Δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Μακμίλαν Σκοτ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο-τρεις προβληματισμούς. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συνοψίσω τα διαμυφθέντα στην συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ, γιατί έχετε ήδη τα κρατά κείμενα και των παρεμβάσεων και των συμπερασμάτων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην λειτουργία και τη νέα, πιο συγκεκριμένα λειτουργία της ΚΟΖΑΚ, ε, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, γιατί αυτή Ζητάμε πιο στενή σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια μέσω ιδίω του ελέγχου της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Αυτό επιφέρει μια περαιτέρω περιπλοκή στις σχέσεις, την οποία πρέπει να μελετήσουμε. Γιατί όπως είπε ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου σε μια συνεδρίαση της διάσκεψης των πρόεδρων, είναι περίπου 400 επιτροπές που έχουν ε, ειδικέ αρμοδιότητες στα πλαίσια των 27 εθνικά κοινοβούλια και περίπου 8.000 οι εθνικοί βουλευτές. να έχουμε λοιπόν σοβαρές σχέσεις με αυτό το πλέγμα ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών εθνικών και εθνικών βουλευτών θέτει πολλά σοβαρά προβλήματα. Ε, τις προάλλες εγκρίναμε μια τροπολογία στην, ε, στον κανονισμό, τροπολογία Μάρτιν, ε, μέσω της οποίας ζητούμε αυτή τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, τη θέλουμε. Και αυτός ο όρος, αυτή η προθεσμία των των 8 εβδομάδων που προβλέπεται αυτή η προθεσμία στο συνοδευτικό πρωτόκολλο της Λισαβόνας ό,τι αφορά την γνωμοδότηση για την επικουρικότητα από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να γίνει πριν από το κλείσιμο, πριν από το πέρας των εργασιών των Επιτροπών. Αυτό σημαίνει πραγματικά περίπλοκες σχέσεις και πολύ έντονη συνεργασία. Τώρα, ποια είναι η λειτουργία της ΚΟΖΑΚ. Ε, η θέση που έχω να πω και για όσα είπε ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ είναι ότι όλες οι ειδικέ επιτροπές θα έχουν μια έντονη σχέση, οργανική σχέση με τις διάφορες, ή με τις δηλαδή διάφορες επιτροπές. Εν τί αυτή περιπτώσει, ε, ποια είναι η λειτουργία της ΚΟΖΑΚ. Είναι να θέσει το θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης όχι μόνο σε επιμέρους ε, νομοθετικές ε, εργασίες και δραστηριότητες. Επομένως, ποιος εκπροσωπεί στο εσωτερικό το, του εκάστοτε Εθνικού Κοινοβουλίου α, και ποιος προωθεί το ευρωπαϊκό συμφέρον. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι πιο αρμόδιες επιτροπές ε, και οι πιο προσκύμενες στην ΚΟΖΑΚ. Χθε με την τροπολογία μας ζητάμε ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής να ηγείται της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΟΖΑΚ. Αυτό είναι ένα θεσμικό μήνυμα που στέλνουμε, ότι η ΚΟΖΑΚ θα πρέπει να έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο και ίσως θα πρέπει να διερωτηθούμε αν η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ΚΟΖΑΚ δεν θα πρέπει να είναι μια ειδική σχέση και να είναι αρμοδιότητα τη επιτροπή μα. Είναι ένα θέμα, ένα πλέγμα από ερωτήματα που θέτω επιτάπητο και δίνω το λόγο για να τα απαντήσει ο, ο αντιπρόεδρος, ο, ο κ. Μακμίλαν Σκότ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η φύση τη εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΚΟΖΑΚ είναι πολύ σημαντική και γνωρίζω πολύ καλά τι συζητήσει που έχουν αναπτυχθεί και στην Επιτροπή σα στο θέμα αυτό. η εμπειρία και η δέσμευση, η στράτευση του Ελμαρ Μπρόκ στη διαδικασία αυτή για την εξέλιξη, για την ανάπτυξη της συνθήκης και στη διάσκεψη, την σταγματική αλλά και μετά, στη συνέλευση νομίζω αλλά και μετά, ασφαλώς του επιτρέπουν να βλέπει με πολύ καθαρό μάτι τα ζητήματα της ισορροπίας ευθυνών και αρμοδιτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Και θα συμφωνήσει πιστεύω μαζί μου ότι η ακρόαση που έλαβε χώρα εδώ πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν έδειξε από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων κάποια πρόθεση η ΚΟΖΑΚ να μετατραπεί σε κάποιο είδου νέα συνέλευση ή κοινοβουλευτικό σώμα. Ασφαλώς βέβαια οι διάφορες αλλαγές που επιφέρει η συνθήκη θα χρειαστούν την, ε, την προσαρμογή ή την διατύπωση μιας νέας μορφής ε, συνεργασίας, πράγμα που επεξεργάζεται ήδη η διάσκεψη των Πρόεδρου, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και άλλα σώματα στο Κοινοβούλιο. Και υπάρχει και μια ομάδα συζήτησης για το, που ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναπτύξει σχέσεις με τα άλλα κοινοβούλια γιατί δεν έχει αρμοδιότητε μόνο η ΑΦΚΟ αλλά και άλλες και υπάρχουν και γκρίζε ζώνε επίσης σε διάφορου τομεί αρμοδιοτήτων. Κύριε Μπρόκ για το όνομα που προτείνω να αλλάξει. Το σκέφτηκα. Ίσως αντί για κόπαρλ να το πούμε κόοπαρλ, δηλαδή ε, συνεργασία, κοινοβούλιο συνεργασία ή συνεργασία κοινοβουλίων και όχι συγκοινοβούλιο. Ως προς την αναγκασόμενη Προεδρία, την κυλιόμενη Προεδρία, πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της ε, μόνιμης Προεδρίας ε, και του, ε, του εκπροσώπου. Ίσως είναι ενδιαφέρον λοιπόν να το δούμε και αυτό. Για τον κύριο Ράγκελ δεν πρέπει να έχει κανένα, δεν έχει κανένα λόγο ανησυχία στο κοινοβούλιο, το εθνικό του κοινοβούλιο είναι από τα πιο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη σχέσεων μέσα από την κόζα του. ως προς τον νέο ρόλο της ΚΟΖΑΚ. Και πάλι στηριζόμαστε σε πληροφορίες, στην ενημέρωση δηλαδή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει όχι μόνο τη γραμματεία αλλά και τα ε, ηλεκτρονικά μέσα υποστήριξης, δηλαδή βάση δεδομένων και τρόπου συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, πρέπει να πω, από όπερες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σπετεριστεί την όλη διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά το Κοινοβούλιο διατηρεί τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όσο δεν αφορά ε, την ερώτηση που έθεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τα χρονικά όρια, που είναι στη τελευταία ανάλυση και κάπως αυθαίρετα, ίσως πρέπει να προσαρμοστούν. Και θα προσαρμοστούν και οι διαδικασίες των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως άλλωστε και η δική μας πρέπει να προσαρμοστεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ανεξαρτήτως των συζητήσεων για τη συνθήκη, η Επιτροπή είχε προσφέρει περισσότερο χρόνο ενημέρωσης και περισσότερη έγκαιρη ενημέρωση ε, το στα κοινοβούλια. Ιδιαίτερα η κυρία Βάλστρομ είχε συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων ενημέρωση. Αλλά δεν είχε ποτέ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ρόλο διαφορετικό από αυτόν που, τις, που προβλέπει η τωρινή συνθήκη. Επίσης λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αναλάβει το βάρος ευθύνη και πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της διαδικασίας. και στην ερώτηση που θέσε ο κύριος Μπρόνς και έτσι αναγκάζομαι να ξαναναφερθώ στο, Ευρω... στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν απαιτείται δηλαδή θεσμικά να γίνει δημοψήφισμα για την έγκριση της συνθήκης, για την κύρωση συνθήκης. Το κόμμα μου μόνο είχε ε, ζητήσει, είχε δεσμευθεί μάλλον ότι αν ε, καταλάβει την κυβέρνηση θα την οργανώσει. Τώρα, όπως είπα, υπαναχώρησε και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Κατά τα άλλα, η διαδικασία όλη για την ε, κύρωση έχει προχωρήσει με απόλυτη ε, νομιμότητα. Κατά τα άλλα, το Κοινοβούλιο έχει διαφορετική θέση πλέον ε, να επιδείξει και χάρη στο νέο καθεστώς των βουλευτών και, και χάρη στο νέο καθεστώς των βοηθών. Και στα 25 χρόνια που έχω εγώ στο Κοινοβούλιο και ο κύριος Μπρόκ επίσης είναι παλιός συνάδελφος, βλέπω ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά και αναβαθμίσει το ρόλο μας και έχω λόγους να σεμνύνομαι γι' αυτό. Αν και, ε, όπως και στο παρελθόν είχα λόγους να ντρέπομαι. Άρα λοιπόν μπορούμε πλέον ε, και να ελέγχουμε τον τρόπο διάθεσης και εκτέλεσης των ε, δαπανών μας και έχουμε μια πολύ αυστηρή νομοθεσία εσωτερική ως προς τον έλεγχο των δαπανών. Δεν έχουμε λόγο λοιπόν να ντρεπόμαστε για τίποτε ή να κρυβόμαστε. Ας προχωρήσουμε και ας εξασφαλίσουμε την σωστή εκπροσώπηση των πολιτών μας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη γενικά για το μέλλον. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κλείνει αυτό το τμήμα της ε, συνεδρίασής μας. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο. Possiamo Με τώρα να επανέλθουμε στην ε, εξέταση του προηγούμενου σημείου, το πέμπτο σημείο της ημεσίας διάταξης, μιλούσε ο εισηγητής, ο κ. Τσασκόφσκι, για το θέμα των ακροάσεων των επιτρόπων. Μιλούσε για τις ερωτήσεις που θα, που θα έπρεπε να θέσουμε στους ε, επιτρόπους. Ο κύριος Σέφη νομίζω ότι είχε μιλήσει και τώρα ποιος άλλος ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Έφνερ. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι στο ερωτηματολόγιο μας δεν θα έχουμε μόνο θέματα ουσίας. αλλά και θέματα που θα μας επιτρέψουν να εξετάσουμε την καταλληλότητα του υποψηφίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ζασκόφσκι για την πολύ καλή προετοιμασία του εγγράφου και κάτι που επισήμανε ο κύριος Ντάφ ίσως δεν ε, αναπτύχθηκε αρκετά στα πέντε αυτά σημεία των προτεραιοτήτων μας. Ήθελα λοιπόν να περιληφθεί αυτό το σημείο στις προτεραιότητες. Αφορά τις σχέσεις μας με τους πολίτες. Άσχετα με το θέμα του εκλογικού νόμου. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας ε, καλό θα ήταν να ενδιαφερθεί για τις ιδέες ε, και τα σχέδια του υποψηφίου επιτρόπου να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η επερχόμενη Επίτροπος Βάλστρομ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό της βελτίωσης της επικοινωνίας με τους πολίτες. Και όποιος και αν είναι ο επόμενος υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει συγκεκριμένα για το τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να βελτιωθούν αυτές οι σχέσεις. Πάντως το έγγραφο είναι πολύ καλό. Απλώς ε, χρήζει κάποιες συμπληρώσει. Σούλτς. Äh, Σας ευχαριστώ. Πολλά ακούσαμε ήδη για το ερωτηματολόγιο και για τις προτεραιότητες. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε κάποιες προτεραιότητες όχι συστάσεις, χρειαζόμαστε περισσότερο προτεραιότητες. Μετά την ε, ψηφοφορία λοιπόν και μετά την ακρόαση με τον υποψήφιο επίτροπο για τα θεσμικά θέματα, θα πρέπει να έχουμε διαμορφώσει γνώμη για το πώς θα προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ιδέα και το ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνημα και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, γιατί υπάρχει μια κόπωση των πολιτών ε, ως προς, ως προς την Ευρώπη. Φάνηκε αυτό και από, την, ε, από το μεγάλο ποσοστό αποχής από τις ευρωεκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε συγκεκριμένα τον Επίτροπο τι σκοπεύει να κάνει για να βελτιωθεί η σχέση της Ευρώπης με τον πολίτη. Τι πρωτοτυπία θα δείξει, τι δημιουργικότητα θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μας με τους πολίτες και αυτή η κόπωση που αισθάνεται ο πολίτης ε, και η μάρα του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεραστεί. Και πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Μπρόκ και στις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και να δούμε πώς ε, θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρξει πρόοδος και όχι παλινδρόμηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια ιεράρχηση και θα πρέπει στην ακρόαση να έχουμε μία βάση για να μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήσεις στον Επίτροπο. Όπως είπε ο κύριος Χέφνερ, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια και η ενημέρωση του πολίτη. Αυτό θα πρέπει να είναι βασικός στόχος της επόμενης Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. κύριος Ράγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Τσουασκόφσκι, ο οποίος ε, προσπάθησε να μας εξηγήσει ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας, όχι μόνο με τις γραπτές ερωτήσεις, αλλά και με τις προφορικές. Συμφωνώ ότι στο σχέδιο προτεραιοτήτων το σημείο υπαριθμών 2 θα πρέπει να πάει στη θέση 1. Φυσικά, ε, το θέμα το, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια πιο ευρεία διατύπωση. Στην προτεραιότητα υπαριθμών 2 εφαρμογή των καινοτομιών που έχει εισαγάγει η συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί νομίζω ότι η προτεραιότητα, προτεραιότητες της Επιτροπής μας τα επόμενα χρόνια θα είναι μια γενική αξιολόγηση της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι είμαστε υπεύθυνοι κατά κάποιον τρόπο για την εφαρμογή ακριβώς αυτή. Πρέπει να δούμε αν τα διάφορα θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς, το Κοινοβούλιο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε τη Λισαβόνα. Νομίζω λοιπόν ότι η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι στο τέλος του 2010 να ετοιμάσουμε μία έκθεση που θα είναι μία γενική αξιολόγηση, μια γενική εκτίμηση όλων των μέτρων που τα διάφορα κοινοτικά θεσμικά όργανα έχουν λάβει, έχουν προωθήσει για να εφαρμόσουν. και να προωθήσουν όλες τις αλλαγές της της Λισαβόνας. Επομένως να την κάνουμε αυτή πρώτη προτεραιότητα και να υποχρεώσουμε και την Επιτροπή που είναι αρμόδια για θεσμικά θέματα να γίνει αρμόδια για αυτή την εφαρμογή. Όπως και εμείς είμαστε για συνταγματικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά που θα κάνουμε αυτά τα επόμενα χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολη ε, αυτή η χρονιά και η Επιτροπή έχει μια έντονη ευθύνη. Εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχουμε την ε, ευθύνη να αξιολογήσουμε και να παρακολουθήσουμε όλα τα τεκτενόμενα σε διάφορα επίπεδα των διαφόρων θεσμικών οργάνων που θα προωθηθούν αυτά τα χρόνια. Θέλω να γίνει αυτή η γενική, εκτίμηση, η γενική αξιολόγηση. Λοιπόν. Κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να περθώ στο σημείο 4 του σχεδίου προτεραιοτήτων. Η ιδέα του ενιαίου εκλογικού συστήματο ε, υποτίθεται ότι θα αυξήσει τη συμμετοχή σε εκλογέ. Λάθο κατά τη γνώμη μου, γιατί η εκτεταμένη αντιπάθεια του πολίτη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οφείλεται στο εκλογικό σύστημα, αλλά στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν πώ θα ψηφίζουν οι πολίτε του και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε είναι πρόβλημα κατά τη γνώμη μου η έλλειψη γνώση του πολίτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ε, ο κόσμος δυσπιστεί απέναντι στην ενημέρωση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα αποφασίστηκε να αυξηθούν τα κονδύλια της ε, ενημερωτική εκστρατεία για τα ωφέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το εγκρίναμε και κάποιος, ο κύριος Φόξ, ο κύριος Μέσσερ Σμιτ, προτάθηκε να δημοσιευθούν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρόταση που καταψηφίστηκε από την Επιτροπή μας. Κατά τη γνώμη μου αυτή η νοοτροπία, αυτή η συμπεριφορά είναι που αποξενώνει και αλωτριώνει τους Ευρωπαίους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το εκλογικό σύστημα. Ευχαριστώ κύριος Μπρόκ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ ιδιαίτερος για τις προτάσεις σας. Μπορούν πιστεύω να αποτελέσουν μια καλή βάση εργασίας. Πριν όμως για διάφορους λόγους θα ήθελα να εκφράσω κάποιες επιφυλάξει προ το εάν η καθολική ψηφοφορία θα πρέπει να αποτελέσει ε, σημείο συζήτησης διότι έχουμε διαφορετικέ παραδόσεις ως προς τα εκλογικά μα συστήματα ως προς την ομοιομορφία, τη στάθμιση κτλ. ανακράτος. Πάντω, έχουμε καταφέρει χάρη συνθήκη του Άμστερνταμ να εισαγάγουμε μία αρχή ενιαία στο εκλογικό μα σύστημα τη αναλογική και αυτό νομίζω προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα στη σύνθεση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό ίσως θα ήταν ε, δύσκολο να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό και άλλων κριτηρίων ή αρχών ως προς το εκλογικό σύστημα γιατί κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε ε, ένα βαθμό μειομορφίας ο οποίος να μην αντιστοιχεί στα, στις παραδόσεις μας. Ε, θα ήθελα πάντως να πω το εξής, ότι εάν, εάν όντως ο πρόεδρος της Επιτροπής προγραμματίζει την σύνθεση της Επιτροπής να την προτείνει κατά τρόπο ώστε να μην είναι ε, δυνατή η έγκαιρη ε, διοργάνωση των ακροάσεων κατά τη διάρκεια του 2009 και χρειαστεί να περάσουμε και στις αρχές του νέου έτους, τότε υπάρχει το εξή πρόβλημα και πρέπει να το καταστήσουμε και σαφές, ότι Ο ύπατος εκπρόσωπος προβλέπει ή τουλάχιστον ακούμε από το Συμβούλιο ότι προβλέπει να αναλάβει τα καθήκοντά του από 1η Ιανουαρίου τουλάχιστον όσον αφορά τα καθήκοντα που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της ε, οργάνωσης όλων αυτών των ακροάσεων θα πρέπει να το καταστήσουμε σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να αναλάβει εν μέρη καθήκοντα η Επιτροπή και δεν είναι δυνατόν να εγκριθεί σε ένα της κομμάτι μόνο η Επιτροπή. Εφόσον πρόκειται να εγκριθεί πρέπει να εγκριθεί και να λάβει καθήκοντα ως σύνολο. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. και ίσως θα ήταν καλό να το ε, διαβιβάσουμε ως τοποθέτηση της Επιτροπής μας, αν φυσικά συμφωνείτε, ε, στην Επιτροπή, έτσι ώστε να προβλέψει αναλόγως ε, τη σύνθεση και τις εργασίες της. Ο κύριος πριν φύγει ο κύριος Μπροκ, θέλω να πω κάτι σημαντικό. Να κάνω μια διευκρίνηση. Να διευκρινίσουμε τη διαδικασία για την ε, υλοποίηση, για την εφαρμογή της ε, συνθήκης. Από 1η Δεκεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη. Και το μέσο ελέγχου, το όργανο ελέγχου, θα κατατεθεί στα πρακτικά ως ο νουπο. Το, για τους Τσέχους, συγγνώμη. Ε, ας με ελέγξει κάποιος Τσέχος συνάδελφος. Επομένως, είμαστε εμπρόθεσμη, ούτω ώστε να, να αρχίσει η συνθήκη να ισχύει από 1η Δεκεμβρίου. Και μπορούμε λοιπόν ε, να έρθουμε σε επαφή με τον υποψήφιο για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικού, όπως και του υπόλοιπους επιτρόπους. Θα υπάρξει επίσημη ακρόαση και θα αποφασίσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και νομίζω θα έπρεπε να μα δοθεί και η επιβεβαίωση ότι έτσι έχουν τα πράγματα στη σημερινή συνεδρίαση. Ο κύριος Γουερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης συνήθως έχουν δύο διακριτές φάσεις. Η έγκριση του συντάγματος, που σε αυτήν την περίπτωση είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, και σε δεύτερη φάση το συνταγματικό κείμενο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δηλαδή, να εφαρμοστούν οι καινοτομίε που περιλαμβάνει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ποια είναι τώρα η ιστορία εδώ, Ότι δεν εξαφανίζονται οι δυσκολίε με την υπογραφή τη συνθήκη και τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη. Γιατί οι διαδικασίε εφαρμογή ε, του κειμένου αυτού που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου ε, είναι διαδικασίες περίπλοκες. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της συνθήκης της Λισαβόνας που δεν θα τεθούν σε εφαρμογή από τον αρμόδιο επίτροπο για συνταγματικές υποθέσεις. Γιατί θα, έχουν, θα είναι αντικείμενο μια ευρείας μεταρρύθμισης της συνθήκες και θα τεθούν σε ισχύ σε διάφορες φάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό προτείνω κάποιες από τις ερωτήσεις που θα κάνουμε στον υποψήφιο για αυτή τη θέση, για αυτό το χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει αυτές τις ίδιες ερωτήσεις να τις θέσουμε και σε υποψήφιους επιτρόπους με άλλα χαρτοφυλάκια, αλλά που έχουν που το χαρτοφυλάκια τους ε, ε, άπτεται του τρόπου εφαρμογής συνθήκης Λισαβόνας. Ε, επομένως, τα σημεία 1 και 2 του ερωτηματολογίου θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε ένα και αυτή η εξωτερική υπηρεσία και οι λειτουργίες του του εκπροσώπου είναι έτη, μια, ε, ακόμα μια ε, συνέπεια της ε, εφαρμογής συνθήκης Λισαβόνας. Σημαντική, αλλά όχι μοναδική. Τώρα, για το ενιαίο ή όχι εκλογικό σύστημα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που αφορούν το εκλογικό σύστημα που θα μπορούσαν να μας αναγκάσουν να τα ξαναδούμε. Παραδείγματος χάρη, αν οι ευρωπαϊκές εκλογές γίνονται την ίδια μέρα σε όλες τις χώρες, αυτό νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή θεώρηση από τους πολίτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε εκλογικούς καταλόγους με υποψήφιους ε, από διαφορετικές εθνικότητες και θα μπορούσαν να γίνουν και μικρές έτσι μεταρρυθμίσεις, με, μικρές εισαγωγές που δεν αλλάζουν την τελευταία απόφαση ε, και τις αρμοδιότητες των εθνικών κρατών, αλλά που αλλάζουν άρδιν την αντίληψη που έχουμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη συμμετοχή, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές εκλογές. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή για να απαντήσει, επειδή νομίζω ότι το καθήκον μου είναι να επαληθεύσω αν υπάρχει δυνατότητα συνένεσης, κατά πλειοψηφία ή δυνατόν για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι, ε, επιτρέψτε μου κύριε Σίγητα, να σας πω, να θέσω το εξή ερώτημα. Υπάρχει ένα θέμα ε, προθεσμίας που έθεσε ο κύριος Νταφ, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι. Είναι η διάσκεψη των Προέδρων το αρμόδιο όργανο θα αποφασίσει. Και με βάση τα νέα που έχουν φτάσει στη γραμματεία, ε, η διάσκεψη των Προέδρων πιστεύει ότι θα τα καταφέρει στο σφιχτόχρονο διάγραμμα. Αλλά θα ξανασυνεδριάσει η διάσκεψη των ε, Προέδρων και θα το θέσουμε αυτό το ερώτημα. Αλλά εμεί δεν είμαστε αρμόδιοι. Εντάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που θα θέσει η δική μα η Επιτροπή, νομίζω ότι βλέπω να σκιαγραφείται μια συνένεση δεν θα πρέπει να κάνουμε δικές μας προτάσεις. Απλώς θα πρέπει να εντοπίσουμε προτεραιότητες. Και σε αυτές θα επιμείνουμε να λάβουμε απαντήσεις από τους υποψήφιους επιτρόπους. Τώρα, για τον έλεγχο θα μας απαντήσει ο κύριος Τσασκόφς. Αλλά σχετίζονται περισσότερο με, το, με την πέμπτη ερώτηση. Τώρα, για τα αρμόδια θέματα, για τα θέματα μάλλον της δικής μας Επιτροπής, ε, θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά όταν εφαρμοστεί η νέα συνθήκη. Σας είπα για την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων, για τη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, ε, για την επιτροπολογία, για την λαϊκή πρωτοβουλία. Προσθέστε και την δική μου πρόταση. Γιατί δεν υπάρχει το εξή στην πρόταση σας, κύριε Σιγητά. Δεν υπάρχει διαδικασία για την προσχώρηση στη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών ελευθεριών. Θα μπορούσαμε λοιπόν και αυτό το στοιχείο να το βάλουμε. Ένα άλλο επίσης, η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το θέμα των επιφυλάξεων που έχουν κάποιες χώρες, ο εκλογικός νόμος, και τη δυνατότητα που έχουμε να ζητήσουμε για νομοθετικές προτάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες βάσει του άρθρου 125. Νομίζω ότι αυτά είπαμε λίγο πολύ. Θα απαντήσει ο κ. Τσασκόφσκι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στη συνένεση. Αφού άκουσα όλους συναδέλφους, πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να διακόψουμε, να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και να εκπονήσουμε ένα κείμενο σε δυο τρει εβδομάδε. Μια και δεν έχουμε το χρόνο για κάτι τέτοιο και δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτού του χρόνου, θα κάνω κάτι συνήθιστο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω, να ανακεφαλαιώσω σύντομα και να υποβάλω και κάποιες προτάσεις, ευελπιστώντα ότι θα καταφέρουμε σήμερα ήδη να καταλήξουμε σε συνένεση λόγω τη πίεση του χρόνου. Θα αρχίσω λοιπόν με το εξή. Πολλοί από εσά, μιλήσατε για την ενημερωτική εκστρατεία προς τους πολίτες, για την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, για τη σύνδεση με τους πολίτες. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σημείο και αντί για το 5 που μιλάει για κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα αναπτύξω ένα θέμα για την επικοινωνία με τον πολίτη που είναι πολύ πιο σημαντικό. Λαμβάνοντας τα σχόλια του Άντριου, του κ. Τσάπλιν και άλλων, και θα συντάξω μία σαφή παράγραφο για την ενημερωτική εκστρατεία, για την σύνδεση της Ευρώπης με τον πολίτη. Νομίζω ότι αυτή είναι μία απλή λύση. ό,τι αφορά την εξέταση του εκλογικού νόμου, είπατε ότι δεν αφισβητήθηκε η σπουδαιότητα αυτού του θέματος, αφισβητείται μόνο η διατύπωση. Γιατί η μελλοντική ομοιομορφία ίσως παρά είναι συγκεκριμένη πρόταση και ίσως επίμαχη. Θα μιλήσω στον, με τον Άντριο, λοιπόν που είναι και ο ειδήμων για τα εκλογικά και θα του ζητήσω να υποβάλει μια νέα διατύπωση για να την εξετάσετε. Θα σας την αποστείλω ήδη από σήμερα τη νέα διατύπωση του Άντριου για το σημείο 4 και μπορούμε άτυπα είτε με τηλεφωνικές συνομιλίες είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να προχωρήσουμε τη συζήτηση και να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο. Άντριου λοιπόν μπορείς να υιοθετήσει μια πιο γενική διατύπωση και ίσως αποφεύγοντας τον όρο ομοιομορφία ή ομοιογένεια, το uniformity, γιατί ο όρος αυτός uniformity είναι πολύ αμφιλεγόμενος. Ας τον παραλείψουμε λοιπόν. Στα σημεία 2 και 1. Συμφωνώ μαζί σας ότι μάλλον θα πρέπει να προταχθεί του 2 έναντι του 1. Και πολλοί το ζήτησαν, γι' αυτό θα αλλάξει σειρά το πρώτο σημείο θα γίνει το σημείο 2 και το σημείο 1 θα ακολουθήσει. Συμφωνώ με τον κύριο Τσόπλιν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάτι πιο γενικό. Να ξεκινήσουμε από τα γενικά. Με το όραμά μας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, αν προτάξουμε την παράγραφο 2, ίσως ε, θα μπορούσαμε να την ε, εμπλουτίσουμε μια πιο γενική πρόταση για το γενικότερο μελλοντικό μας όραμα και όχι με τις λεπτομέρειες και θα έχουμε ούτως ή άλλως ε, την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψει του Επιτρόπου για τα θέματα αυτά γιατί υπάρχουν πολλέ ε, γενικές ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο και ο Επίτροπος ή η Επίτροπος θα αναπτύξει τις ιδέες του για το ρόλο του, τις προτεραιότητές του κτλ. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με δύο λόγια, δύο λόγια για το μελλοντικό όραμα της Ένωση. Επίσης θα πούμε δύο λόγια και για τη γενική αξιολόγηση. Μια-δύο τέτοιε γενικέ λοιπόν προτάσει και μετά θα επισέλθουμε στι λεπτομέρειε τη εφαρμογή. Το δεύτερο σημείο θα είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, το θέμα της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνθήκης, αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό που αξίζει μια χωριστής παραγράφου. Η πρώτη παράγραφος λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα είναι ουσιαστικά η δεύτερη από εμά, αλλά θα περιλαμβάνει και μια γενικότερη πρόταση για το όραμα του Επιτρόπου για το μέλλον, για τις συνθήκες, επίσης ε, μια γενική αξιολόγηση και μετά θα μιλούμε για τις λεπτομέρειες τη εφαρμογή της συνθήκη Λισαβόνα. Αυτή θα είναι η πρώτη παράγραφο. Η δεύτερη παράγραφο θα αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Η τρίτη παράγραφο θα μιλάει για την ενημερωτική εκστρατεία και την σύνδεση και επικοινωνία με τον πολίτη. Αυτή την παράγραφο θα την εκπονήσω σήμερα με τη βοήθεια του Άντρη, όπως είπα προηγουμένω. Και σημείο 4, ε, Στοκχόλμη, σημείο 5, εξέταση του εκλογικού νόμου. Εκεί θα υποβάλει μια εναλλακτική διατύπωση ο Άντριου. Θα τα συντάξω λοιπόν όλα αυτά σε λίγο. Θα σας τα στείλω ηλεκτρονικά. Και όποιος θέλει να μου επισημάνει κάτι, να μου τηλεφωνήσει, να μου στείλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε σήμερα, αύριο, να φτάσουμε σε νέα συνένεση που ελπίζω ότι θα ανταποκρίνεται στις ε, στην κρατούσα θέση της Επιτροπής, γιατί δυστυχώς χρόνο για μια νέα συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση δεν έχουμε, όπως ε, μου υπενθυμίζει η Γραμματεία. Πάντως, ήδη αν από τώρα έχετε σχόλια για τις τελευταίες μου προτάσεις, ε, να τα συζητήσουμε. Βέβαια, αναφέρθηκαν και άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Ο πρόεδρος επισήμανε ένα τέτοιο. Την ε, προσχώρησή μας στην ε, συνθήκη ανθρωπίνων, στη, χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης ο κύριος Ιγουάρεγκη μίλησε για τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις αυτοεξαιρέσεις και τι, γίνεται, θα γίνει στο μέλλον ή για την προσχώρηση της Κροατίας. Νομίζω ότι θα γίνει ό,τι συνέβη και στις προηγούμενες ε, διευρύνσεις. Όταν τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται το ευρώ, έχουν δυνατότητα αυτοεξαίρεσης. Ε, τα νέα κράτη-μέλη όμως που θα προσετεριστούν το ευρώ δεν μπορούν να, έχουν, να τύχουν αυτοεξαίρεση. Είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν του ε, ισχύοντες κανόνε. Και δεν πρόκειται να εξετάσουν το θέμα, να συζητήσουν το θέμα του ευρώ. Το ίδιο θα ισχύσει και για την Κροατία και τις ε, ε, υποψήφιες χώρες ω προς το χάρτη. Θα πρέπει δηλαδή οι νέες χώρες τις διαπραγματεύσεις να δεχθούν ε, όλους τους κανόνες. Δεν θα έχουν τέτοια δυνατότητα αυτοεξαίρεση όπω όπως η Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία και η Τσεχία για τη χάρτα θεμελίδα δικαιωμάτων. Άλλωστε το θέμα αυτό που ε, αναφέρθηκε είχε μάλλον συμβολικό χαρακτήρα. Αυτά τα πρωτόκολλα ούτως ή άλλως μερικές φορές έχουν ε, έχουν περισσότερο διακοσμητικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα είναι αρκετά για να διαμορφώσουμε γνώμη για τον Επίτροπο. Πάντως ε, και στην ακρόση θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλες ερωτήσεις. Αυτό που είναι σημαντικό, γιατί για την απάντηση όλων αυτών των ερωτήσεων θα είναι προετοιμασμένος ο Επίτροπος. Θα έχει χρόνο να τις εξετάσει, να ετοιμάσει ωραίες φράσεις ε, και γλαφυρές. Το θέμα είναι εμείς ε, αυθόρμητα να υποβάλουμε μερικές ε, νέες ερωτήσεις για να δούμε πώς αντιδράσει ο Επίτροπος εκείνη τη στιγμή. Και επίσης θα δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις του στις γενικές ερωτήσεις. Εκεί που θα αναπτύξει το γενικό του όραμα για την Ένωση, για τις θεσμικές ή διοργανικές σχέσεις, για τις προτεραιότητές του. Για πολλά θέματα ο υποψήφιος ή υποψήφια επίτροπος θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όχι μόνο την περιέργειά μας, αλλά και τις προσδοκίες μας για το μέλλον της Ένωσης. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε και αυθόρμητες προφορικές ερωτήσεις που θα γίνουν θερμό για να δούμε πραγματικά πώς και ο Επίτροπος είναι έτοιμος αυθόρμητα να απαντήσει και πώς θα απαντήσει ενστικτοδός, χωρίς την προετοιμασία που θα προϋποθέτει η απάντηση στο ερωτηματολόγιο. Αυτά συνοπτικά. Υπήρχαν και πολλά άλλα σημαντικά σχόλια, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όχι χρόνο, αλλά χώρο για να τα συμπεριλάβουμε ανασυντάξω λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες. Αν έχετε ήδη σχόλια ή προτάσεις, πολύ ευχαρίστως να τις ακούσουμε. Και θα τις λάβω υπόψη τις επόμενες ώρες που θα εκπονήσω τις πέντε νέες ερωτήσεις με τις προτεραιότητές μας. Μάλιστα, νομίζω όντως υπάρχει μια συνένεση για την πρόταση του εισηγητή του κ. Τσασκόφσκι. Ναι, από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, όχι με τυπικό τρόπο, αλλά ουσιαστικό τρόπο, γιατί πραγματικά θαύμασα την ακρίβειά του και τη σοβαρότητα με την οποία ανέλαβε αυτό το συμμετείχε στη συζήτηση. Τελειώσαμε στην πράξη. Τι μένει, μόνο να αποφασίσουμε την ημερομηνία της νέας συνεδρίασης. Θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου από τις 15 ε, μέχρι 18.30 και την 30 ε, Δεκεμβρίου αυτό, έτσι, η Δευτέρα και 3η 1 1η Δεκεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30. Επίσης, ε, Λίμπε Γιούρι και εμείς θα συνεδριάσουμε από κοινού για να ψηφίσουμε την, το ψήφισμα για το πρόγραμμα Στοχόλμη. Στοχόλμης. Θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου, προσεχώς, δηλαδή πολύ προσεχώς, από τις 2 μέχρι τις 3 στις Βρυξέλλες. Αυτά ευχαριστώ.